Mes chers collègues, bonjour. Καλησπέρα σα. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά. Παρακαλώ πολύ, είστε λίγο θορυβόδης σήμερα. Ε, τις ευχές μου για το καινούριο χρόνο. Ε, μακάρι να σας φέρει υγεία, ευτυχία και επιτυχία σε όλα σας τα εγχειρήματα και κυρίως τα εγχειρήματα στο εσωτερικό της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Υιοθέτηση ημερήσιας διάταξης. Υιοθετούμε την ημερήσια διάταξη χωρίς αντιρρήσεις. Ωραία. Δεν έχω να κάνω ανακοινώσει. Θα ξεκινήσω με το πακέτο κινητικότητα για τις χερσαίες μεταφορές με τους εισηγητές μας, την κυρία Ντεμπονφουά, την κυρία Κλούν και τον κύριο Σαλίνη. Συνάλφοι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας για ένα σύνολο νομοθετικών προτάξεων σχετικών με τις χερσαίες μεταφορές. Το πακέτο δηλαδή κινητικότητα 1, όπως το λέμε εμείς, στο ιδιόγλωσσό μας. Πολύ σημαντική αυτή η δουλειά γιατί σχετίζεται με την ζωή δεκάτων χιλιάδων επαγγελματιών του κλάδου καθώς επίσης και με την ανταγωνιστικότητα χιλιάδων επιχειρήσεων μεταφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη μας λοιπόν είναι μεγάλη εναντί όλων αυτών. Πέραν όμω των πτυχών αυτών που είναι ιδιαίτερα σημαντικέ, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις σχετικές με την κινητικότητα και το περιβάλλον. η υγεία των πολιτών μα, οι εκπομπές ρήπων, η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, στο πώς θα οργανώσουμε την κινητικότητα στις χερσαίες μεταφορές ε, και στο συνδυασμό μεταφορών. Ευθύνη λοιπόν μεγάλη για μας. Και πρέπει να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Για να υιοθετηθεί μια ε, νομοθεσία κατάλληλη και προσαρμοσμένες ανάγκες ε, θα πρέπει να ακούσουμε ένα τον άλλο, και να σκεφτόμαστε τις απόψεις των υπολείπων προς όφελος των πολιτών μας και των επαγγελματιών του κλάδου. Σας λέω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας ε, να αποφασίσουμε με βάση κομματικές γραμμές. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Σε ό,τι αφορά την διοργάνωση των ορασιών, θα ξεκινήσουμε να εξετάσουμε, εξετάσουμε μια πρόταση ε, πρώτες προς πρόταση. Καταρχήν θα δίνω το λόγο στον εισηγητή, μετά στους και εισηγητές, κατόπιν στους βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο, κατόπιν στον εισηγητή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τον οποίο καλωσορίζω, και στην Κομισιόν. Τη συζήτηση θα κλείνει κάθε φορά ο εισηγητής θα ξεκινήσουμε με την οδηγία Ευρωβινιέτας και την κυρία Ρεβό Νταλόν, Μπονφουά, που είναι η συγγήτρια. Μετά θα περάσουμε στην πρόταση για την φορολόγηση των οχημάτων, με συγγήτρια την κυρία Κλούν. Καλώς ήρθατε. Και τέλος θα περάσουμε στην οδηγία για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων διοδίων με εισηγητή τον κύριο Σαλίνη. Έχουμε ένα συνολικό χρόνο, τον οποίο έχουμε καθορίσει για, το, για τις τρεις αυτές προτάσεις. Παρακαλώ πολύ να είσαστε λοιπόν προσεκτικοί. Με το χρόνο σας θα είμαι αυστηρή, διότι θέλουμε οι τρεις αυτές προτάσεις να συζητηθούν εξίσου, όχι μία εις βάρος της άλλης. Δίνω λοιπόν το λόγο καταρχήν στον κύριο Κούλο, πρόεδρο του Τμήματος Μεταφορών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό να μας ε, πείτε συνοπτικά ε, ε, την άποψή σας για την συνεργασία μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για ένα θέμα όπως αυτό δεν μπορούμε να προφανώς να αγνοήσουμε ένα μέλος, ε, ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της. Είτε πρόκειται για την Κομισιόν, είτε πρόκειται για τους εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών, είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλοι μαζί θα πρέπει να συνεργαστούμε αρμονικά σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό όπως είπατε και εσείς διότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία απαραίτητη ως ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το περιβάλλον που είναι η ζωή δική μας και το παιδιών μας αύριο. Και τρίτον, τα εκατομμύρια των εργαζομένων που χρειάζονται καλές συνθήκες εργασίας. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε καλέσει. Σήμερα είναι μια πρώτη επαφή αυτή. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους πολίτες της. Ξεκινάμε δυναμικά, κύριε Κουλόν. Μπράβο. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρεβόνταλόν, μετά στους και ηγητές και στα άλλα μέλη που θέλουν να πάρουν το λόγο. Κυρία Ρεβόνταλόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση της έκθεσής μου, θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση, αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα το κείμενο να αναβαπτιστεί ε, οδηγία Eurocharging ή Euro ε, ευρωτέλη στα ελληνικά. Ε, εμείς θέλουμε να βγούμε από ένα σύστημα ευρωβινιέτας. Ε, ο τίτλος αυτός νομίζω ότι παραπλανά λοιπόν αυτή η πρότασή μου δεν αποτελεί ακρογωνίο λίθο βέβαια <laughs> της εκθεσής μου, αλλά πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να υιοθετηθεί. Αν η οδηγία ευρωτελών ε, επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα αποφεύγει τις τρευλώσεις ε, και τις διακρίσεις, ε, ε, δεν αποτελεί από μόνη της το εργαλείο για την υλοποίηση της Λευκής Βίβλου και του κανόνα ορυπένων πληρώνει. Όπως σας είπα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια καλή πρόταση. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή σε όλα τα ε, βαρέ οχήματα, η συμπερίληψη των ελαφρών οχημάτων, ε, η, η σταδιακή απαγόρευση της Ευρωβινιέτας, η δυνατότητα προσαυξήσεων λόγω συμφόρησης, ε, η δυνατότητα λήψης υπόψη των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι προτάσεις που βοηθούν να λάβουμε υπόψη την πραγματική χρήση των υποδομών ε, και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν δεν έφτασε μέχρι το άκρο της λογικής αυτής. Καταρχήν, προτείνει ένα σύστημα ε, καταργής της βινιέτας χωρίς Όμω, ε, απαραίτητα να αντικατασταθεί το σύστημα με σύστημα τέλων. Δεύτερον, η Κομισιόν προτείνει την συμπερίληψη των ελαφρών οχημάτων στο πεδίο εφαρμογή, ε, επιτρέπει διακρίσει ανάλογα τι κατηγορίες οχημάτων. Υπ' αυτή την έννοια, προτείνω καταρχήν όχι μόνο να απαγορεύσουμε τις βινιέτες για τα βαρέα οχήματα, αλλά να τις αντικαταστήσουμε με τέλη που θα ε, υπολογίζονται με βάση την ε, απόσταση. Μετά το τέλος της ε, χρήσης των μηνιατών το 2006 για τα ελαφρά οχήματα προτείνω επίσης και εκεί την χρήση επιβολή τελών σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Δηλαδή από 1η Ιανουαρίου 2026 τα τέλη να εφαρμόζονται όχι μόνο στα ε, βαρέα οχήματα αλλά και στα ελαφρά οχήματα και στις μοτοσυκλέτες. Η εφαρμογή αυτών των τελών βέβαια θα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Αυτή είναι μια ε, φιλόδοξη πρόταση αλλά απαραίτητη αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με το στόχο της εξάλληψης των διακρίσεων και προκειμένου να εφαρμόσουμε πλήρως την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτής της αρχής, προτείνω να εισάγουμε ένα τέλος εξωτερικών δαπανών για όλα όσα καλύπτονται ε, από ε, τέλος υποδομών. Και από το 2026 και μετά αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα. Παράλληλα με την εφαρμογή των δύο αρχών, ο χρήστη πληρώνει και ο ρηπαίνων πληρώνει, η διαφάνεια των συστημάτων διοδίων ε, αποτελεί σημαντικό στόχο στις προτάσεις μου. Για να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτά αυτά τα συστήματα προτείνω τα εξή. Πιστεύω ότι Αν εισάγουμε μία... Ε, αν, αν τέλη ε, που θα σχετίζονται με τη χρήση ε, των υποδομών ε, θα γίνουν πιο εύκολα δεκτά τα διόδια. Επίσης προτείνω εκπτώσεις 13-50% σε χρήστες οι οποίοι έχουν κοινωνικές ανάγκες βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου, απομακρυσμένες κλπ. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την εδαφική συνοχή, προτείνω να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη ή στις τοπικές αρμόδιες αρχές για να λαμβάνουν υπόψη κάθε φορά ε, τον αντίκτυπο των διοδίων στις ε, ε, πιο απομακρυσμένες περιοχές και στις περιφέρειες. επίσης, τα, διόδια θα πρέπει να δαπανώνται εκεί που συλλέχθηκαν και εισπράχθηκαν. Τέλος, για να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτά τα διόδια για, από τους μεταφορείς, ε, εισάγω στο κείμενο την υποχρέωση ύπαρξης πάρκινγκ ασφαλών ε, ε, χώρων στάθμευσης κατά μήκο των οδικών αξώνων. Επίσης, ο διαχειριστής της ε, υποδομής θα πρέπει ε, να διαφημίζει τη χρήση των ε, διοδίων που εισπράττονται και των τελών. Δεύτερον, ε, μία ανεξάρτητη αρχή ε, θα, ε, εποπτείας θα πρέπει να ασχολείται με την χρήση των λαπανών και με την διαφάνεια των διοδίων. τέλος θα μπορούσε αυτό να είναι και ένα καθήκον μιας Ευρωπαϊκής Αρχής. Έχω και άλλα μέτρα που προτείνω στην έκθεσή μου για να απλοποιηθεί το σύστημα ε, προς ε, καθώς επίσης και για την απλοποίηση της γραφειοκρατίας προκειμένου να μην βαραίνει υπερβολικά τους χρήστες. Προτείνω επίσης να δοθεί η δυνατότητα ε, των ε, ε, δαπανών. θα ήθελα να δείτε τις προτάσεις αυτές στο σύνολό τους, σαν ένα σύνολο. Μόνο έτσι θα καταλάβετε την πλήρη, τους, την πλήρη αξία των προτάσεών μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι, όσοι ε, ήρθαν σε επαφή μαζί μου, μα ξέφρασαν την άποψή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν, με την οποία συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά. Τον Σαμιουέλ Μπελέ, τον ε, βοηθό μου δηλαδή, και τον ε, βοηθό της ομάδας. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και περιμένω να ακούσω και τη δική σας άποψη των σκιωδών εισηγητών καταρχήν και των υπολείπων μελών της Επιτροπής μετά. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame Σας ευχαριστώ κυρία Ρεβόνταλον. Ξεκινάει η συζήτηση λοιπόν. Θα ξεκινήσω με τους σκιώδεις εισηγητές. Τρία λεπτά ο πρώτος σκιώδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω <clears throat> την εισηγήτριά μας για την εξαιρετική δουλειά την οποία έκανε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η τροποποίηση του τίτλου είναι ιδιαίτερα έγκυρη σαν πρόταση, γιατί εξακολουθούμε να μιλάμε για ροβινιέτ ενώ το σύστημα αυτό θέλουμε να το καταργήσουμε. Μετά από τις συζητήσεις ε, για τη Λευκή Βίβλο των Μεταφορών καταλήξαμε σε συγκεκριμένες θέσεις σχετικά με την εφαρμογή της αρχής ε, του «Όποιος μολύνει πληρώνει». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε την ε, λογική μας και έκανε μια πρόταση η οποία γενικά είναι ισορροπημένη και ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Λυπάμαι όμως γιατί ούτε η εισηγήτρια ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξεφράστησαν σαφώς υπέρ μιας δεσμευτικής και στοχευμένης χρήσης των πόρων που θα προέλθουν από τις δραστηριότητες αυτές. Τώρα για την έκθεση της Κριστίνα. Να πω ότι είναι μια φιλόδοξη έκθεση, μια θαραλέα έκθεση. Σε ορισμένα σημεία μου δημιουργεί την εντύπωση ότι <clears throat> αποκλίνει το πλαισίου το οποίο θα πρέπει στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα βρούμε μια ισορροπημένη συμβιβαστική πρόταση. Υπάρχει ένα θέμα, είναι η λήψη υπόψη και των δευτερευουσών οδικών συστημάτων ε, ε, οδών. Εδώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Νομίζω ότι αν κάποιο έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει το δευτερεύον οδικό δίκτυο για να αποφύγει την επιβολή των διοδίων, είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει ε, κάποια προβλήματα, πρέπει να συζητηθεί. Η πρόταση της εισηγητρίας για τη λήψη υπόψη και των οικολογικών παραγόντων ε, με κάνει να αναρωτηθώ με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ποια είναι η μέθοδος και τώρα και η έκπτωση 50% για τους τακτικούς χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το, το δικό σύστημα για να μεταβούν στο χώρο εργασίας τους είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και αυτό αντικείμενο συζήτησης περαιτέρω για να αποφύγουμε κάποια φαινόμενα γραφειοκρατικής δυσανάλογα υψηλής επιβάρυνσης. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις και όχι να προσθέσουμε προβλήματα. Το θέμα τώρα της φορολογίας των βαρέων οχημάτων ανάλογα με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και γι' αυτό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφώς ε, ε, ε, περισσότερο ρεαλιστική. Πάντως, <clears throat> θα πρέπει όλες, ε, για λόγους συνοχής, όλοι οι τρόποι μεταφοράς να τύχουν υποστήριξης. Η συμπερίληψη τώρα των λεωφορείων, ε, τουριστικών λεωφορείων, αλλά ακόμα και των διτρόχων, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. σχετικά τώρα με τα μικρά φορτηγά τα οποία κάνουν τις διανομές και αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί συζητήσεις. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τους μικρούς μεταφορείς και για την διανομή προϊόντων και πακέτων. Οι μεταφορείς αυτοί δεν θα πρέπει να υποστούν πλήγματα στο επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους. θεωρούμε παράλληλα ότι η συμπερίληψη ε, του κόστους των ατυχημάτων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί θέμα. Όπως επίσης και οι θέσεις ε, του συναδέλφου της ε, CESE e για μεγαλύτερη διαφάνεια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε. Και νομίζω ότι η συγγήτρια κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση απαιτείται στα κράτη-μέλη οι προτάσεις των πολιτών να ληφθούν υπόψη. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα συνεργασία, ευχαριστώ και για τη μέλουσα συνεργασία. Η πρόεδρο βιάζεται όμως και σταματώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπάρ. Κοιτάξτε, δεν είμαι και πολύ αυστηρή, σας έδωσα δύο επιπλέον λεπτά, μην με κατηγορείτε ότι είμαι αυστηρή. Ο κύριος Βαντάλεν, τρία λεπτά έχει το λόγο. Θα τα καταφέρετε. Καλησπέρα Πρόεδρε. Να <clears throat> σας καλησπερίσω όλους. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα θα ήθελα να πω ότι Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες ακόμα ε, στα πλαίσια της διατύπωσης της έκθεσης αυτής. Η συζήτηση στην πολιτική μου ομάδα συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί. Σέβομαι μέχρι κάποιο σημείο τις φιλοδοξίες της εισηγήτριας πάντως. Η διεύρυνση της εμβέλειας του πεδίου εφαρμογής έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και τα δίκυκλα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερο σοφό. Ένα άλλο σημείο στο οποίο έχω κάποιες επιφυλάξεις είναι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των χρηστών και να εξαρτηθεί η επιβάρυνση από την οικονομική κατάσταση των χρηστών. Έχω αμφιβολίες γι' αυτό. Σκεφτείτε να μπούμε σε μια τέτοια λογική χωρίς τέλος. Και τώρα μια ειδική ευρωπαϊκή αρχή για τις οδικές μεταφορές δεν την επιθυμούμε όπως επίσης και απορρίπτουμε ε, και την φορολόγηση ή καλύτερα την επιβολή διοδίων ε, για την χρήση των ε, δικτύων δευτέρου επίπεδου, των οδικών δικτύων δευτέρου επίπεδου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια σωστή βάση υπολογισμού για, τον, για τα διόδια και φυσικά η αρχή του όποιος μολύνει πληρώνει είναι μια βασική αρχή και θα πρέπει να εφαρμοστεί σχετικά τώρα με την προσημείωση σε εισαγωγικά των εσόδων από τα διόδια αυτά. Είναι καλή ιδέα να συνδεθούν τα ε, έσοδα των διοδίων, ε, αλλά εδώ βρίσκεται το θέμα της αρχής της επικουρικότητας και εδώ δεν θα πρέπει να προκαταλάβουμε κάτι. Πάντως αυτό το οποίο με ικανοποιεί είναι ότι η συγγήτρια λέει ότι εκεί όπου εφαρμόζονται ε, συγκεκριμένες επιβαρύνσεις ε, θα πρέπει να υπάρχουν και ε, σταθμοί ε, στάθμευσης, μάλλον χώροι στάθμευσης ασφαλής για τους οδηγούς γιατί κινδυνεύουν δυστυχώς πολύ συχνά οι οδηγοί των μεγάλων οχημάτων από παραβατικές συμπεριφορές στους χώρους στάθμευσης σήμερα. Φυλασσόμενα πάρκινγκ λοιπόν είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Η συγγήτρια λέει ότι θα πρέπει να δώσουμε ε, ειδική μεταχείριση, να επιφυλάξουμε ειδική μεταχείριση για τα οχήματα τα οποία μολύνουν λιγότερο. Θα συμφωνήσω μαζί της, η συζήτηση και στην ομάδα μου συνεχίζεται και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρία λεπτά και ούτε ένα δευτερόλεπτο παραπάνω. Πετύχατε λοιπόν τον στόχο σας. Ο κύριος Τέλιτσκα έχει το λόγο. Για τρία λεπτά. Ο κύριος Μακρόν επισκέφτεται τη Βόρεια Γαλλία σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτή την πρόταση, αλλά γι' αυτό λόγο το Ντομινίκ Κρικέ δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα, οπότε θα παρουσιάσω εγώ τα σχόλια. Θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω εμείς βέβαια στην ομάδα μας, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ποιες θα είναι οι απόψεις μας, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για την ποιότητα της έκθεσής της. Η πρόταση Κομισιόν βαίνει προς σωστή κατεύθυνση και η έκθεση της κυρίας Ρεβό Νταλόν βελτιώνει ακόμα περισσότερο την πρόταση Κομισιόν. Ε, υποστηρίζουμε την, ε, τα διόδια ε, που θα βασίζονται στην γεννηθήσα απόσταση ανάλογα με την κατηγορία, κατηγορία του οχήματος και σύμφωνα με την αρχή του ο πληρώνει και ο, ε, ο χρήστης πληρώνει. Το ίδιο συμφωνούμε και με τον στόχο τα ποσά που εισπράττονται από τα διόδια να κατανοούνται σε συγκεκριμένες δράσεις που θα έχουν σχέση ε, με την συντηρήση των υποδομών ε, ή την ε, πρόθεση της εισπράξης των διοδίων κλπ. Επίσης στηρίζουμε την εισηγήτρια ε, στην πρόταση δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Χερσαίων Μεταφορών. Θα θέλαμε βέβαια να δούμε κάποιες διευκρινήσεις, για παράδειγμα, ότι γίνεται αν υπάρχουν ε, ήδη εκχωρήσεις στη διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων ή ποιος θα είναι αρμόδιος για την απόφαση της εφαρμογής των διοδίων στο δίκτυο. Τέλος, η τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν ε, οι αρμόδιες αρχές, κάθε αρμόδια περιφερειακή αρχή να μπορεί να επιβάλλει ε, διόδια στην επικράτειά της. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ. Και εγώ προέρχομαι από την ίδια περιφέρεια που, θα ήταν, που είναι ο κ. Ρικέ, αλλά προτίμησα να είμαι εδώ μαζί σας και όχι με τον πρόεδρό μας. Οπότε είστε τυχεροί που είμαι εδώ. Ah, c'est M. Dalunde qui prend la parole. Excusez-moi. M. Dalunde, la parole est à vous. Thank you, Madam Κύριος Dalunde. Έχει πολλές θετικές πτυχές αυτή η πρόταση κομισιόν το δεδομένο για παράδειγμα ότι καλύπτει όλα τα οχήματα, ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση τη διανθήσα απόσταση κλπ. Όμως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ο, τον υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα στους διάφορους τρόπους μεταφορών και θα πρέπει να δούμε τα τέλη στα οχήματα ε, μαζί με τα τέλη στις δρομικές μεταφορές και να τα συγκρίνουμε για να μην δημιουργούνται διακρίσεις. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στους βουλευτές που δεν είναι σκιώδεις ηγητές. Ένα λεπτό ο καθένας. Κυρία Φώστερ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και είναι πολύ γενναιόδωρο ο χρόνο που μου δίνεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγητρία για τα σχόλια που έκανε. Δεν μιλάω εξ τη ομάδα. Προφανώ προφανώς ε, μιλάω προσωπικά από πλευρά τη αντιπροσωπείας μου. Δεν μας ε, ενοχλεί από πλευρά της Ευρωπητροπή που θέλουμε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή. Δεν υποστηρίζουμε να, τη συμπερίληψη των λεωφορείων, των ε, πούλμαν και σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση της ζωής των ανθρώπων που ζουν στην Ήπετρο. Διαφωνούμε με την ε, αξίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η κατηγορία γυρολάς είναι πλέον ε, παροχημένη και σε ό,τι αφορά τις προτέρα Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι οι... υπάρχουν σωστές ή ποσοστοί υπολογισμοί για τις ε, εκπομπές και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την αρχή του ορίου πένων πληρώνει, σύμφωνοι, αλλά θα πρέπει να αποφασίζει κάθε κράτος μέλος το πώς ε, επιβάλλει τέλη βάση χρόνου, για παράδειγμα, γιατί πιστεύουμε ότι το δικό μας σύστημα ε, λειτουργεί και δεν θέλουμε να επιβληθούν περιπλοκές αλλάζοντα το. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την επιβολή των τελών αυτών, αυτό και πάλι αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών και νομίζω ότι τέλο πάντων καταλάβατε το πνεύμα μου. Δεν έχω τίποτα προσωπικό κατά τη εισηγήτρια, αλλά ε, μα, είναι οι άποψει μα αυτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φώστερ. Και είδατε ότι σα έδωσα και 30 δευτερόλεπτα παραπάνω. Πολύ ευγενικό εκ μέρου μου. Ε, κυρία Αρνοτού. Merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Θα επανέλθω στην ουσία, το δεν θα επανέλθω μάλλον στο περιεχόμενο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να σχολιάσω λίγο τις προτάσεις της κυρίας Σανταλών που είναι απαράδεκτες. Ε, οι αστικές μεταφορές δεν θα πρέπει να τύχουν μιασδήποτε μορφής ε, ε, <clears throat> φορολογίας για οποιονδήποτε λόγο. όπως επίσης και η αποκλειστική χρήση των εσόδων στην τοπική ε, ζώνη στην οποία εισπράττονται είναι μη πρακτικό και απαράδεκτο θέμα που δεν την αρχή της επικουρικότητας. Λέγει η έκθεση ότι η φορολογία των φορτηγών και των βαρέων οχημάτων ε, αλλά και η φορολογία των μοτοσυκλετών σαν παράδειγμα είναι κάτι το εντελώς απαράδεκτο λόγω των υψηλών φόρων που ήδη πληρώνουμε για τα καύσιμα. Σχετικά τώρα με τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, να θυμίσω ότι οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στην δημιουργία μιας κοινωνικής ανταγωνιστικής ζούγκλας. Δεν θέλουμε λοιπόν μια τέτοια πρόταση. Η κυρία Ιάλα Σέντερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για τις προτάσεις της. Πολλές από αυτές είναι ενδιαφέρουσες. Η τροπολογία 56 όμως προτείνει ένα σύστημα για να βοηθήσουμε τις ε, περιφερειακές χώρες όπως η Ισπανία. Όμως, να σας πω το εξής. Θα προτιμούσαμε να είναι ευρωπαϊκό μέτρο, όχι περιφερειακό. Γιατί ξέρουμε πως ε, τα ε, κράτη-μέλη πάντοτε προσπαθούν ε, να επιβάλλουν τέλη υπόλοιποι, αλλά όχι να μην επιβάλλουν τέλη στους δικούς πολίτες. Επίσης διαφωνούμε με, τις, με τα διόδια στα περίχωρα πόλεων, διότι τις πιο φτωχέ οικογένειε, τις έχουμε τελικά στείλει εκεί και τώρα να του βάλουμε και διόδια στις μετακινήσεις του νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Τρίτον, η ανεξάρτητη αρχή ε, σε εθνικό επίπεδο λέει η συγγήτρια για να μην γίνουν διακρίσεις όμως ενδεχομένως θα ήταν καλύτερο η αρχή αυτή να είναι ευρωπαϊκή. Τέλος, ε, η η ανάλωση των εσόδων σε συγκεκριμένους σκοπούς ίσως είναι καλή πρόταση, αλλά δυστυχώς σε ορισμένες χώρες το Σύνταγμα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όπως στην Ισπανία, ε, όλα τα έσοδα πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών και από εκεί διατίθενται. Επίσης, η τροπολογία 49 και 50 θα ήθελα να αλλάξουμε το κείμενο το σχετικό με τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Δεν καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό. Το βγάζουμε από την πρόταση Κομισιόν και το βάζουμε κάπου αλλού. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική πίσω από αυτέ τι τροπολογίε 49 και 50. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την εισηγητρία. Νομίζω ότι προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται σε ό,τι αφορά τα έσοδα, ε, το earmarking των εσόδων. Ε, ναι, κατά πόσον ε, ε, τώρα πώς θα, θα διαμορφωθεί το θέμα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ τα δύο για παράδειγμα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει επικουρικότητα. Για παράδειγμα, ύστερα το κόστος ε, για τη συμφόρηση. Πιστεύω ότι απλά πρόκειται για ένα τέλος και νομίζω ότι κανείς δεν προκαλεί μα, σκόπιμα συμφόρηση για την εφαρμογή. Θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν διασυνοριακά και ομοιόμορφα για να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό βάση χρόνου και όχι βάσει απόστασης, ε, συμφωνούμε. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερος μέθοδος. Merci, Madame à vous. Κύριε Ντεμόντε. Ευχαριστώ. Καταρχάς ξεκινώντας να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους Σκιώδης σχετικά τώρα με το τέλος ε, che hanno destato una resistenza iniziale ma poi sono stati accettati eh, dai σχετικά με το τέλος συμφόρησης νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να επιβαρύνει απευθείας τους πολίτες σχετικά τώρα με τις τροφολογίες οι οποίες έχουν προταθεί η αναφορά που γίνεται για το δευτερεύον οδικό δίκτυο είναι κάτι το οποίο προκαλεί την προσοχή μας, γιατί τα δίκτυα αυτά είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα, είναι μια μορφή διαμετακόμισης η οποία ελαφρύνει πολλές φορές τους αυτοκινητοδρόμους και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα μόλυνσης. Επίσης είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση που γίνεται για τους χώρους στάθμευσης. Και σχετικά με τα διόδια θα ήθελα να πω ότι τα διόδια για την χρήση υποδομών θα πρέπει τα έσοδα να επενδύονται ακριβώς στην διαχείριση και τον, την βελτίωση των ίδιων των υποδομών. Η αρχή φυσικά του όποιος μολύνει πληρώνει φυσικά, αλλά από την άλλη με σταδιακό τρόπο γιατί θα μπορούσαμε να βρούμε και κάποια αντικίνητρα υπέρ των σιδηροδρόμων σε αυτή την περίπτωση. Ε, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε κυρία Ιγιούτο. Είστε σκιώδης εισηγήτρια. Έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ε, το αεροπλάνο μου καθυστέρησε. Και συγγνώμη και για τη φωνή που είναι βραχνιασμένη. Σχετικά λοιπόν με το συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε τέσσερα βασικά σημεία πάνω στα οποία έχουμε ήδη εκφράσει τις θέσεις μας οι οποίες περιλαμβάνονται στις προτάσεις που έγιναν σχετικά με, τις, με το κόστος των υποδομών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, βρίσκω ότι είναι θετική η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας είναι και αυτό ε, θετικό ε, και η αύξηση επίσης ε, του πεδίου επιβολής και στα λεωφορεία και τα μικρά λεωφορεία, τα μίνιμπας. Η επένδυση στην συντήρηση των υποδομών είναι πολύ σημαντικό θέμα με το οποίο συμφωνούμε. Με τα λεγόμενα εξωτερικά κόστη ε, το θέμα της χρήσης ε, της δυνατότητας συμπερίληψης των εξωτερικών μορφών κόστους, δηλαδή βλάβες στο περιβάλλον κτλ. Πρέπει να είναι μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τη χρήση μέσων τα οποία να μην μολύνουν. Τα κόστη αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη μείωση της μόλυνσης. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την ίδια λογική που χρησιμοποιούμε και για τα κόστη ε, που καλύπτουν τις υποδομές. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ε, στόχοι οι οποίοι να είναι άμεσα αποσβέσιμοι. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν για την ε, καταπολέμηση της μόλυνσης, για την διάδοση εναλλακτικών μορφών μεταφορών που δεν μολύνουν, έτσι ώστε να δημιουργηθούν υποδομές για να αναπτυχθεί η αγορά αυτή η οποία δεν έχει βοηθηθεί διόλου ε, και να μπορέσουμε να μετακινηθούμε και σε άλλες μορφές μεταφορών και για τους επιβάτες έτσι ώστε να περάσουν από το αυτοκίνητο στο τρένο και το ίδιο να ισχύσει και για τα εμπορεύματα. Να ξεφύγουμε λοιπόν από τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων αλλά να περάσουμε σε άλλες μορφές πιο αβιώσιμες οικολογικά και αηφόρες σχετικά με το κόστος του τέλους συμφόρησης. Καλό είναι να εφαρμοστεί. Από την άλλη όμως και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική επιβολή κόστους ε, μεταφορών και σε άλλες μορφές μεταφορών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα τελευταίο σημείο σχετικά με την διαφάνεια. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει, ε, να ξεκαθαρίσουμε το τι θέλουμε ακριβώς και για ποια κόστη μιλάμε. Δηλαδή κόστη διαχείρισης, κόστη υποδομών και εξωτερικά κόστη θα πρέπει να δούμε τι πλεονεκτήματα μπορούμε να έχουμε σε σχέση με την χρήση αυτών των μεθόδων. Ε, τι μείωση έχουμε σε επίπεδο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ε, τι ωφέλη έχουμε χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά ε, σε επίπεδο αποσυμφόρησης των οδικών δικτύων. Ποια είναι η πιθανή μείωση των ατυχημάτων και ποια τα κέρδη σε επίπεδο ασφαλείας. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά σημεία στα οποία θα κρίνουμε το πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Γιούτο. Στρέφομαι τώρα στον εισηγητή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Δίνω το λόγο στον κύριο Ματσόλα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση για να σας παρουσιάσουμε την άποψη της ε, Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα χρησιμεύσει και ε, για τη μείωση των εκπομπών. Εμείς θεωρούμε ότι η οθέτηση ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης ε, και επιβολής διοδίων ανάλογα με τα χιλιόμετρα ενός συστήματος μη γραφειοκρατικού και λαμβάνοντας υπόψη και τα εξωτερικά κόστη για όλες τις μορφές οχημάτων και η εφαρμογή επίσης της αρχής όποιος μολύνει και όποιος χρησιμοποιεί πληρώνει είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την βελτίωση και την αποσυμφόρηση των οδικών δικτύων. Στους όρους αυτούς τους οποίους προανέφερα, εμείς πιστεύουμε σαν Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή ότι το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά και στα βαρέα οχήματα και στα ελαφρά οχήματα και με προτεραιότητα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Η Επιτροπή βλέπει με ανησυχία ότι απαιτούνται 130 δις κατέτος σε επίπεδο επενδύσεων σε, στην Ευρώπη ε, και είναι δυστυχώς ε, τα διαθέσιμα χρήματα πολύ λιγότερα από ό,τι πριν από την αρχή της ε, κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν τα χρήματα τα οποία θα εισπράττονται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη, την συντήρηση ε, και την σωστή εκμετάλλευση των ε, μέσων υποδομών που δημιουργούνται. Θα πρέπει να μειώσουμε την στροφή προς τις οδικές μεταφορές, να βελτιώσουμε τους τρόπους λειτουργίας των σιδηροδρόμων, να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε από την αυτοματοποιημένη οδήγηση. Απαιτείται ευελιξία ιδιαίτερα για τις περιφερειακές περιοχές, τις ορεινές περιοχές και τις νησιωτικές περιοχές. Θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα μέτρα αυτά και να τα οικειοποιηθούν οι χρήστες και οι καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπέρ της σωστής και ξεκάθαρης ενημέρωσης για το πώς θα χρησιμοποιούνται τα έσοδα και πώς θα επενδύονται τμήματα των εσόδων αυτών. Απαιτείται να υπάρξουν ε, σύνθετοι δείκτες των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει επίσης ε, να δημιουργηθούν και θέσεις απασχόλησης από τις πολιτικές αυτές. Εμείς θέλουμε να ελέγχονται και οι επιστημονικές βάσεις τεκμηρίωσης της οδηγίας και με βάση τις εμπειρίες ε, του Μπρένερο ε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε και σε επίπεδο διασταυρώμενης χρηματοδότησης. Η μοναδική παρατήρηση την οποία κάνουμε στην πρόταση της εισηγήτριας αφορά την εσωτερική αγορά. Κατά τα άλλα να συγχαρώ την εισηγήτρια και την προσοχή την οποία έδειξε στη δική μας έκθεση στην πρότασή της περιλαμβάνει πολλές από τις προτάσεις μας. Την ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ κύριε Ματσόλα. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τις ευχές σας, τις έχουμε ανάγκη φέτος. Νομίζω ότι θα είμαι εύκολος ε, για αυτή την έκθεση και ευχάριστος εισαγωγικά, γιατί εμείς δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε την πρόταση αυτή. Συγχαίρουμε άλλωστε την εισηγήτρια για την ποιότητά της, που επιβεβαιώνει ε, τις βασικές αρχές ιδιαίτερα σε ορισμένα θέματα όπως το εξωτερικό κόστος. Η κυρία Ρεβόντα Λόν πηγαίνει πέραν των προτάσεων της Επιτροπής για την εφαρμογή της αρχής ομολύνων πληρώνει. Δεν θα σταθώ τώρα σε όλες τις κατατεθήσεις τροπολογίες, αλλά να αναφερθώ σε κάποιες που θεωρούμε πιο σημαντικές. Καταρχάς, η διεύρυνση της εμβέλειας της οδηγίας είναι βασική ε, και στη δική μας αρχική πρόταση. Άκουσα κάποιες επιφυλάξεις από ορισμένους συναδέλφους σας σχετικά με τη διεύρυνση στα λεωφορεία, ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε προβλήματα σε ένα μέσο δημόσιας μετακίνησης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να εξαιρέσουμε τα λεωφορεία από τα διόδια, γιατί χρησιμοποιούν τις υποδομές. Ε, επίσης υπάρχει και το phasing out, το σταδιακό του συστήματος των βινιέτ, μετά από μια βατική περίοδο να περάσουμε σε συστήματα διοδίων, στα οποία η Επίτροπος επιμένει. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να κάνω αναφορά είναι η κατανομή των πόρων, των εσόδων, το earmarking ε, εμείς θα συμφωνήσουμε με αυτό, αν και πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί, γιατί ε, πρέπει να μάθουμε από αυτά τα οποία ζήσαμε μέχρι τώρα και από τις φαλιάρες που φάγαμε από τα κράτη-μέλη, αλλά παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρουσα η πρότασή σας και είμαστε υπέρ, ιδιαίτερα υπέρ των τροπολογιών που προτείνει η συγγήτρια. Να σημειώσω τρία επιμέρους σημεία πάνω στα οποία η συζήτηση θα πρέπει να συνεχιστεί. Το πρώτο σημείο είναι η αρχή της ουσιαστικής μεταρρύθμισης των διοδίων. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε σχέση με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης, μεταρρύθμισης και ανακοίνωσης από πλευράς των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δίνει την τελική αδειοδότηση πριν τροποποιήσουμε την πρόταση αυτή απαιτείται λίγη προσοχή γιατί αυτές οι υποχρεωτικές ανακοινώσεις από πλευράς των κρατών μελών έχασαν ή μάλλον απέδειξαν την αξία τους γιατί επέτρεψαν ένα διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι τα διόδια ήταν απαραίτητα και συμβατά με την οδηγία. Τώρα, οι επιστροφές τις οποίες ή μάλλον οι εκπτώσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 50% στους τακτικούς χρήστες. Αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκω υπερβολικό και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο της τιμολόγησης που είναι κυρίως η μείωση της συμφόρησης. Βέβαια αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να συνδυάσουμε τους διαφορετικούς στόχους και να λάβουμε υπόψη μας στόχους σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο εδαφικής συνοχής. Είναι μια τροπολογία αυτή όμως την οποία θα πρέπει να εργαστούμε ακόμα περισσότερο. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις φιλοδοξίες της κυρίας Ρεβόντα Λόν σε επίπεδο εξωτερικού κόστους. Ίσως εδώ κάτι το ελάσσον πάνω στα οποία θα πρέπει να σταθούμε επιφυλακτικοί είναι η συμπερίληψη των τελών των προερχόμενων και του κόστους από ατυχήματα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί όταν διαβάζει τις μελέτες γύρω από τα θέματα αυτά. Τελειώνω με ένα θετικό τρόπο να σημειώσω την τροπολογία 35. Στην τροπολογία αυτή ε, η συγγήτρια μας λέγει ότι στα οδικά δίκτυα στα οποία υπάρχουν διόδια πρέπει να υπάρχουν ποιοτικέ υποδομές και πρέπει να υπάρχουν χώροι στάθμευσης ε, ασφαλούς Νομίζω ότι είναι μια τροπολογία αυτή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία σαφώς και δικαιολογεί αν θέλετε την κωδικοποίηση εφόσον πληρώνει ο α, έχει δικαίωμα σε ποιοτικέ υποδομές όχι μόνο στο δρόμο αλλά και στις περιοχές στάθμευσης, στους χώρους στάθμευσης. Και αν υπάρχει μια τροπολογία η οποία αποδεικνύει τις σχέσεις αυτές είναι μια τροπολογία η οποία αποδεικνύει ότι με τις εκθέσεις που θα συζητηθούν και αύριο έχουμε ένα συνολικό πακέτο οδικών μεταφορών. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τις κοινωνικές πλευρές και τις πλευρές της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και συνδέονται οι κοινωνικές πλευρές με τις πλευρές τιμολόγησης των, ε, της χρήσης των υποδομών. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ρεβόντα Λόν, θα σας ξαναδώσω το λόγο για 1,5 λεπτό. Αλλά βλέπετε ότι όλοι σας στηρίζουν, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστημένη είναι. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους σας για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Τα σημειώνω όλα. Έτσι κι αλλιώς τώρα ξεκινάμε. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα σχόλια που έγιναν. Το θέμα των προσαυξήσεων το ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι. Κάποιοι ανυπομονούν κιόλα. Ευχαριστώ πολύ και την στήριξη της Κομισιόν και την Κομισιόν μάλλον για τη στήριξή της. υποχρεωτική διάθεση σε συγκεκριμένα έργα ε, μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρη στο κείμενο. Υπάρχει ήδη, μπορούμε να την διευκρινίσουμε. Ε, δεν ξέρω τι υπήρχε στο, τι, ποιες ήταν οι δυσκολίες στο παρελθόν να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό από τα κράτη-μέλη. Αλλά πάντως πιστεύω ότι αν υιοθετήσουμε αυτή την, ε, αυτή την πρόταση θα γίνουν πιο εύκολα δεκτά τα τέλη. Τώρα, ε, η εσωτερικοποίηση δεν είναι... Ε, συγγνώμη, η, τα διόδια σε, δε, δε, σε μικρότερους δρόμους και οδούς είναι προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά. Προσφέρουμε απλώς τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, πολύ σημαντικοί, μίλησε η κυρία Γιάλα Σέντερ γι' αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα τα, τα, στα κράτη-μέλη να μην γίνονται διακρίσεις για αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να πάρουν συγκεκριμένου δρόμους για να πάνε στο σπίτι τους. Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, αναφέρθηκε ότι δεν λαμβάνω υπόψη επαρκώς ε, τις ε, χαμηλές εκπομπές ορισμένων οχημάτων σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του ύψους των διοδίων. Δεν είναι αλήθεια αυτό, αλλά αν μπορώ να βελτιώσω το κείμενο, πολύ ευχαριστώ. Εγώ λέω ότι μπορεί να γίνει και έκπτωση 75% για αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών. Ε, αυτό εξυπηρετούν και οι τροπολογίε 49 και 50, κυρία Γιάλα Σέντερ, για να διευκρινίσω δηλαδή τα πράγματα. Πρόκειται για τροπολογίες διευκρινιστικές όχι για να αποσύρω την πρόταση της Κομισιόν ή να την καταργήσω. Σε ό,τι αφορά και πάλι την υποχρεωτική διάθεση σε συγκεκριμένα έργα, ε, αντιλαμβάνουμε ότι έχει πολύ υποστήριξη αυτή η πρόταση. Θα πρέπει όμως να πείσουμε και αυτούς οι οποίοι δεν είναι ακόμα ε, σύμφωνοι. Θα πρέπει βέβαια να λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορετικές χρήσεις των υποδομών. Προφανώς όταν ένα, ένα όχημα είναι καθαρό θα λαμβάνεται υπόψη. Τέλος, 20 ε, ε, Φεβρουαρίου ε, η υποβολή των τροπολογιών 19 με, 14 και 15 Μαΐου η απόφαση στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Μας αναφέρατε και το ε, χρονοδιάγραμμα. Θα σας το πω και εγώ. Ε, τροπολογίες υποβάλλονται, υποβάλλονται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα θα το δούμε. Ωραία. Και περνάμε στον, στην επόμενη συγκεκριτήρα, την κυρία Κλούν, για την φορολόγηση των οχημάτων. Κυρία Κλούν, έχετε το λόγο θα ακολουθήσουν οι σκιώδεις ηγητές και τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι αυτό το θέμα συνδέεται με το προηγούμενο, αλλά ε, ουσιαστικά αφορά κάποιου όρου ό,τι αφορά την φορολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα κράτη-μέλη να έχουν πιο μεγάλο πεδίο εφαρμογή για να, μειώσουν, να μειώσουν του ε, συντελεστέ ε, φορολόγηση κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα που είχαν οριστεί με την οδηγία για την Ευρωβινιέτα. Γενικά λοιπόν η Επιτροπή μας συμφωνεί με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να πω προφανώς αυτή εξ αρχή ότι η φορολόγηση αποτελεί θέμα και αρμοδιότητα των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπό διαβούλευση. Το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη προφανώ και τι απόψει του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή, αλλά δεν δεσμεύεται από την απόψη του Κοινοβουλίου, γιατί προφανώ υπάρχει η αρποκλειστική αρμοδιότητα. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Καλώ ορίζουμε ωστόσο τι προτάσει για να ανταποκριθούμε σε κάποιε από τι προτάσει ε, για τι οδικέ μεταφορέ σε ό,τι αφορά κοινωνικό, οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπημένη προσέγγιση που να αναγνωρίζει και τη σημασία των οδικών μεταφορών για τη λειτουργία τη ενιαία αγορά. Και πιστεύω προσωπικά ότι αυτή η επιβολή τελών βάση απόστασης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ισότητα και πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι σε ό,τι αφορά την εισαγωγή των μέτρων αυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε περίπτωση οι εθνικές ιδιαιτερότητε και θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία για τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά ενδεχόμενο διοικητικό κόστος το οποίο ενδεχομένως να θεωρηθεί άδικο και επιβαρυντικό για τον τομέα των μεταφορών. Εισαγάγοντα, λοιπόν, αν εισαγάγουμε ε, φορολόγηση βάση απόστασης, θα πρέπει να μειωθεί η φορολόγηση για να περιοριστεί και η επιβάρυνση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως. Είναι σημαντικό επίσης να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση διπλής επιβολής ε, τελών αυτό είναι άλλωστε και ο στόχος της πρότασης αυτής. Είμαι υπέρ λοιπόν της μείωσης ε, του φορολογικού συντολιστή σε επίπεδο για περίοδο 5 ετών και θα πρέπει να υπάρχει και εδώ κάποια ευελεξία για να απλοποιηθεί κάπως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μην αποτελέσει ενδεχόμενο διοικητικό κόστος για τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό στην πρότασή μου, στις ε, τροπολογίες μου, προτείνω να μειωθεί το επίπεδο φορολόγησης σε ένα βήμα και όχι σταδιακά, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πέντε στάδια. Το πιο σημαντικό σημείο, ωστόσο, είναι ότι εδώ μιλάμε για διαβούλευση στο θέμα αυτό. Και φυσικά σε συνάρτηση και με το προηγούμενο θέμα το οποίο συζητήσαμε, προσβλέπω στα σχόλια και τις παρεμβάσεις των συναδέλφων προκειμένου να ολοκληρώσουμε, ελπίζω, το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Του. Από τους σοσιαλιστές, μάλλον, το λόγο έχει ο κύριος Έρτουκ τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ και καταρχά θα πρέπει να σα πω ότι αντικαθιστώ την συνάδελφό μου την Κλόντια, η οποία δυστυχώ δεν μπορεί να παραβρεθεί εδώ σήμερα. Η κυρία Ταπαντέλη λοιπόν τοποθετείται ως εξής. Η... Ο υπολογισμό βάσει τη απόσταση μπορεί να δώσει μεγάλο κίνητρο για τη μετάβαση σε μια καθαρή οικονομία μεταφορών. Καλωσορίζουμε λοιπόν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ την κατεύθυνση αυτή. Και η κυρία Τιμπαντέλη συμφωνεί ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ υποστήριξη των ε, επενδύσεων σε υποδομέ, μείωση τη συγχωρήπανση ε, και τη περιβαλλοντική ρήπανση και στην παρούσα φάση τα τρέχοντα οχήματα δεν αποτυπώνουν την πραγματική χρήση, ενώ τα διόδια θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια λύση για το μέλλον. Ωστόσο, ανακύπτουν δύο ζητήματα τα οποία θα ήθελε να τονίσει για να πετύχουμε μια ισόρροπη προσέγγιση στο θέμα αυτό. Καταρχάς, η μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολόγησης για τα οχήματα, για τα AGV, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον υπάρχει ένα σύστημα επιβολής φορολόγησης βάση απόστασης για να μην υπάρχει διπλή φορολόγηση αλλά να μην υπάρχουν και ανισορροπίες για τις τοπικούς και εθνικούς προϋπολογισμούς γιατί κάποιες χώρες ε, εξαρτώνται από τα έσοδα των φόρων και, και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά την ε, περίοδο για τη μείωση αυτή πιστεύει ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το πώς θα επηρεάσει αυτό τις εκάστοτε κυβερνήσεις η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει η μετάβαση αυτή σε πέντε έτη αποτελεί πρόβλημα για τα θεσμικά εκείνα όργανα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν και την νομοθεσία τους, να ενημερώσουν την νομοθεσία τους. Και καλωσορίζει λοιπόν τις αλλαγές της κυρίας Κούν. Κλούν. Ε, και το να γίνει αυτό σε δύο-τρία στάδια θα ήταν πιο διαχειρίσιμο. Σας ευχαριστώ κυρία Κλούν για τη δουλειά που κάνατε και η κυρία Ταμπαρντέλ προσβλέπει στη συνεργασία για να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ την εισαγωγή ε, της ε, υπολογισμού βάση απόσταση και του χρονικού πλαισίου στο οποίο θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγέ αυτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρε. Ο κύριο Βαντάλαν έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Συγγήτρια. Συμφωνούμε με αυτά που λέει ότι θα πρέπει να δώσουμε πιο πολύ ευελιξία στα κρατημέλη για τη μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή γιατί θα πρέπει να αφήσουμε και ελεύθερη την περίοδο μέχρι το 2024 και αυτό αποτελεί ένα θέμα το οποίο συζητιέται στην ομάδα. Ξεκινήσαμε να το συζητάμε, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά φυσικά η ευελιξία πάντα είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνα το ECR. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Φαντάλαν. Ο κύριος Ρικέ, ποιος τον αντικαθιστά. Η κυρία Πελπάο, θα πάρει το λόγο. Α, η κυρία Μάισνερ. Έχει το λόγο. Όχι, όχι, δεν μου έδωσε κάποιο κείμενο. Δεν ξέρω ποιος θα τον αντικαταστήσει. Απλά θα πρέπει ενδεχομένω να μην τον αντικαταστήσει κανείς. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Δεν θα ακούσουμε λοιπόν την παρέμβαση του κυρίου Ρικέ. Η κυρία Μακάρθη έχει τώρα το λόγο. Δεν είναι παρούσα. Ο κύριος Ντάλλοντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και οι φόροι και τα τέλη θα μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ επικοδομητικό εργαλείο για να δώσουμε κίνητρα στους καταναλωτές για την αγορά πιο σωστών οχημάτων. Και εκ παραλληλού δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στη ρυθμίση των τελών. Το θέμα είναι και η αγορά των οχήματων. Και εδώ θεωρώ ότι τα κίνητρα ψυχολογικά παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι καταναλωτές έχουν την επιλογή σε ό,τι αφορά το όχημα δηλαδή που επιλέγουν και ως τώρα δεν είχε τόσο μεγάλο ρόλο η κατανάλωση. Βασικό κριτήριο ήταν το κόστος αγοράς. όσοι εκπέμπουν πιο, πολύ καυσαέρια, πιο πολλά καυσαέρια θα πρέπει πολύ απλά να πληρώνουν πιο πολλά από όσου είναι πιο καθαροί σε τα οχήματά του. Και αυτό προφανώ θα αποτελέσει κίνητρο. Θα πρέπει να λεφθεί υπόψη λοιπόν αυτό ως ε, στοιχείο καλή και επιβολή τελών και φορολογία, αλλά και το θέμα της αγοράς των οχημάτων είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ και τώρα εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Λεσβάκη πάλι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω και εγώ λοιπόν με την ίδια δόση αισιοδοξία. Υποστηρίζω λοιπόν την έκθεση της εισηγήτριας της κυρίας Κλούν η οποία συμφωνεί με τη βασική πρόταση της Επιτροπής να υπάρξει ευελιξία στα κράτη-μέλη για τη μείωση των φορολογιών στα φορτηγά και να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη να, ξεκίσουν, ξεφύγουν από το σύστημα το φορολογικό και να περάσουν σε ένα ε, σύστημα επιβολής τελών. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό για τα κρατη Το τονίζουμε. Είναι η ευελιξία αυτή που θα υπάρχει στο μέλλον. Υπάρχει μία τροπολογία στο σχέδιο της έκθεσης που θεωρούμε ε, ότι απλοποιεί παραπάνω το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντί για πέντε στάδια προβλέπονται ένα στάδιο η εισηγητρία προτείνει να γίνει αυτό ένα έτος με μόνο μία φάση. Γιατί όχι. Αλλά αν περάσει αυτή η τροπολογία, γιατί να υπάρχει αυτό το επίπεδο αυτή η μεταβατική φάση για τη μείωση της φορολόγησης μέχρι το 2024. Θα μπορούσε να γίνει αυτό πολύ νωρίτερα στην περίπτωση αυτή, εφόσον υπάρχει μόνο ένα στάδιο. Και η ημερομηνία θέση σα εφαρμογή τη αναφερμένη οδηγία. Αυτό είναι το μόνο το οποίο ήθελα να αναφέρω. Και πάλι όμω επαναλαμβάνω για μια έκθεση την οποία στο σύνολό τη καλωσορίζουμε ιδιαίτερω. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Και έτσι αισιόδοξο σα θέλω γιατί έχουμε και άλλη μια έκθεση. Η κυρία Μάισνερ Βρήκετε την τοποθέτηση του κυρίου Ρικέ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ναι, ενημερώθηκα μόλι ότι το έγγραφο του κυρίου Ρικέ αφορά και τι δύο εκθέσει. Το άφησε εδώ η συνάδελφο. Να σα πω λοιπόν ότι ο κύριο Ρικέ ευχαριστεί και την ε, κυρία Κλούν για την έκθεση αυτή, η οποία κινείται προς σωστή κατεύθυνση και υποστηρίζει το σύστημα επιβολής ιδιών με βάση την απόσταση, το οποίο φαίνεται ότι συνάντη με την αρχή του ορυπενών καθώς και την ε, συμπεριλήψη των εξωτερικών τέτοιων παραγόντων. Γι' αυτό λοιπόν και υποστηρίζει και τις διεκθέσεις, τις τροπολογίες που θα θέλει να διευκρινίσει, με τις τροπολογίες του μάλλον και θα ήθελε να διευκρινίσει κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα του ποιο θα είναι αρμόδιος για να αποφασίσει για τα τέλη και την επιβολή διαδίων. Και τέλος, ε, τίθεται και το θέμα ε, της επιβολής διαδίων και τελών σε επίπεδο υποεθνικό, σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό. Γι' αυτό λοιπόν δεν έδωσα κάτι ξεχωριστό για την έκθεση αυτή, καθότι το, η παρέμβαση ισχύει και για τι διεκθέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μάιστερ και τώρα το λόγο πάλι έχει η συγγετρία, η κυρία Κλούν, για να κλείσει. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ και για τα μέλη και την Επιτροπή που, για τι παρεμβάσει του. Και νομίζω ότι και πάλι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συμφωνία για την εισαγωγή σε επιβολή διοδίων με βάση την απόσταση. Θα πρέπει να γίνει αυτό με τρόπο μείωσης της ε, επιβολής ε, φορολόγηση στα οχήματα και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν υπάρχει προφανώς υποχρέωση για τα κράτη-μέλη για κάτι τέτοιο. Πρόκειται για κατευθυντήριε γραμμές. Είναι σημαντικό προφανώς να αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο της φορολόγησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις. Και να αναγνωρίζουμε ότι ασφαλώς αν αυξηθεί κάπου η φορολόγηση, θα πρέπει να μειωθεί κάπου αλλού για να μην υπάρχει άδικο συναγωνισμό, αθέμητο συναγωνισμό. Θα συνεχίσω τη συνεργασία με του σκιώδει σε περίπτωση που υπάρξουν τροπολογίε του επόμενου μήνε. Και είμαι βέβαιη ότι θα μα ενημερώσετε και για τι προθεσμίε και για το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρο, σωστά τα λέτε. Άρα, για τροπολογιών, προθεσμία 20 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι. 20 Φεβρουαρίου. Και συμφωνήσουμε λοιπόν με την έκθεση για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων διοδίων. Και το λέγω, έχει ο κύριος Σελήνη, καλώς ορίσατε και χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. Να ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή και μετά τους κοιόδες εισηγητές και έχουμε και ε, πάλι έναν εισηγητή από την Ευρωπαϊκή και Οικονομική Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Um, il η έκθεση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα τι διόδια είναι κάτι το οποίο οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η οδηγία του 2004 δεν εφαρμόζεται πλέον. Οι βασικές ανησυχίες άπτονται κυρίως του κεντρικού θέματος της διαλειτουργικότητας των συστημάτων διοδίων ηλεκτρονικών διοδίων, όπως επίσης ε, υπάρχει τίθεται και το θέμα της ανταλλαγής ε, πληροφοριών διαμεθοριακού τύπου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, των, ε, το πρόβλημα της μη πληρωμής διοδίων από διάφορες κατηγορίες και χώρες. Νομίζω ότι αυτή είναι η στοχή τους οποίου έχουμε. Βασικό στόχος είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο από τη μία θα παρέχει ε, μια υπηρεσία με βάση ένα συγκεκριμένο μηχανισμό, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει να προσέρχονται σε διάλογο ουσιαστικά όλα τα συστήματα των κρατών μελών. Υπάρχουν σήμερα όρια και περιορισμοί. Υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια πρόσβασης στην αγορά σε σχέση με την παροχή της συγκεκριμένη υπηρεσίας. Επιβάλλονται ε, βαρύς φόροι σήμερα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πάνω στο οποίο θα πρέπει να παρέμβουμε. Ένα δεύτερο θέμα αφορά το κόστος των μηχανισμών. Σαν παράδειγμα το δορυφορικό δίκτυο ε, ο στόχος προς τον οποίο κινούμε θα είναι αυτό σήμερα και το κόστος του είναι πάρα πολύ υψηλό. Θα πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε τη συμβίωση των διαφορετικών μηχανισμών με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην προκληθεί ανυπόφορο ύψος κόστους. Έχουμε επίσης και το θέμα του συσχετισμού με τα συστήματα εφιούς μεταφοράς. Έχουμε προβλήματα επίσης ε, σύμπτωσης των συχνοτήτων. Υπάρχει θέμα νομικής βάσης επίσης που οδηγεί σε ελλείψεις στις πληρωμές. Συνολικά θα έλεγα λοιπόν ότι ο ε, ε, εισηγητής κάνω κάποιες προτάσεις τις οποίες έχω ήδη θέσει υπόψη και στους κοιόδης ιδιαίτερα στις πιθανές συνέργειες που μπορεί να υπάρξουν με τα συστήματα των ευφυών μεταφορών. Δεν θα συμφωνήσουμε με την ιδέα τροποποίησης της συχνότητας των τηλεδιοδίων, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε πάρα πολύ ψηλά παράδεκτα κόστη. Δεν μπορούμε να πάμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Ε, νομίζω επίσης ένα βασικό θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση σήμερα είναι η ανάγκη, η χρήση των, των τεχνολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται αντίθετα με την προηγούμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενταχθεί στο κυρίως κείμενο και όχι σε προσάρτηση του κειμένου. Συνολικά λοιπόν η ανησυχία μας έγινε κυρίως στην διατήρηση της συνοχής με την οδηγία Ε, Υπάρχουν διαφορές στους ορισμούς ε, του τι είναι ελαφρύ όχημα σαν παράδειγμα. Πρέπει εδώ να υπάρξει μεγαλύτερη συμβατότητα. Ε, πρέπει να υπάρξουν ε, κάποιες τροποποιήσεις που θα οδηγήσουν σε σωστή κατανομή των ρόλων των διαφορετικών επιπέδων. Θα αποκλείσουμε στα πλαίσια ε, των τηλεδιοδίων ε, κάποιες άλλες ε, ιδέες ανάγνωσης των πινακίδων κυκλοφορίας. Είναι ένα σύστημα το οποίο νομίζω ότι ναι μεν λειτουργεί εν μέρη αλλά δεν είναι αξιόπιστο. Δύο τελικές παρατηρήσεις σχετικά με την επιβολή, το enforcement. Δεν έχουμε εδώ κάποιες συγκεκριμένες διαφορές αλλά κάποιες διευκρινήσεις θα θέλαμε Προτείνουμε μια αναθεώρηση κάποιων σημείων του κειμένου σχετικά με τα εθνικά σημεία επαφής. Ε, τα εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να θέτουν στην συγκεκριμένη κρατική υπηρεσία της τράπεζας δεδομένων τις οποίες έχουν όπου δεν έχει γίνει μία πληρωμή. Ε, πάντως συνεργαζόμαστε σωστά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θέλουμε ε, να δούμε ακριβώς το πού θα καταλήξει η εργασία της ομάδας εργασίας για τα ηλεκτρονικά διόδια και νομίζω ότι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσουμε την συνεργασία έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις που θα μεταφερθούν στη νέα οδηγία. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω το, τη συζήτηση αμέσω. Δίνω καταρχήν το λόγο στην κυρία Σενάλοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή, κύριο Σαλίνη. Δεν έχω και πολλά να πω, κυρίως να συμφωνήσω μετά όσα ανέφερε. Δεν επιθυμώ την ενοποίηση στα 5,9 GHz όλων των ηλεκτρονικών διοδίων. Η, επίσης, η, τεχνολο... η αλλαγή των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, θα πρέπει να μπορεί να γίνει μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε συνεργασία. Επίσης, θα ήθελα να δούμε το έργο της Επιτροπής για τα Διόδια και αν ε, η μελέτη τους ε, μας λύει έγκαιρα θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε με την οδηγία και να συμπεριλάβουμε για κάποιους οδηγούς από τη μελέτη στην οδηγία στο άρθρο 2. Και κάποιε άλλε τροπολογίε θα ήθελα να σχολιάσω. Η οδηγία, για παράδειγμα, θα έπρεπε να καλύπτει και ε, διόδια για την είσοδο στις, ε, ε, στο κέντρο των πόλεων ή σε περιοχές χαμηλών εκπομπών. Υπάρχουν χώρες οι οποίες εισάγουν διόδια για την είσοδο στο κέντρο. Είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση. Περιμένω να συνεργαστούμε με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σενάλοβα. Ο λόγος στον κύριο Δεμέρσμεκερ. Ο κύριος Τόσενόφσκι, σκιώδης ηγητής μας, δυστυχώς ε, λείπει, ζητά συγγνώμη, οπότε παίρνω εγώ τη θέση του. Θα σας παρουσιάσω τις απόψεις του για την έκθεση του κύριου Σαλίνη. Ως και ο συγητής μας πιστεύει ότι η έκθεση αυτή είναι ισορροπημένη. Στηρίζουμε ιδιαίτερο στην τροπολογία παριθμών 6, έτσι ώστε ο κατάλογος των τεχνολογιών να παραμείνει στη διαδικασία συναπόφασης και όχι με κατεξιοδότηση πράξη όπως προτείνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Είσαστε πραγματικά συνοπτικότατος. Ο κύριος Βαν Εγώ θα μιλήσω λίγο παραπάνω όντω. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για την σχέδια έκθεση και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η λειτουργικότητα των συστημάτων διοδίων θα πρέπει να πραγματευτεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και όπως ξέρετε υπάρχουν διάφορα πάθυρακια τα οποία τελικά όμως ε, Μα παρεμποδίζουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επιβάλλει την πρότασή τη και θα πρέπει να δούμε πώ θα εγγυηθούμε τη λειτουργικότητα των συστημάτων αυτών με την πρόταση αυτή σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τη μη καταβολή διοδίων στην Ένωση γιατί θα πρέπει να ελέγχεται πιο εύκολα και αυτό θα προωθήσει τελικά την ενιαία αγορά και φυσικά τώρα ωφελούνται όσο δεν πληρώνουν. Χρειάζονται λοιπόν καθαροί και ξεκάθαροι κανόνε για την ε, καταχώρηση, για την επιβολή διοδίων και φυσικά θα πρέπει να διατηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα πρόστιμα σε περίπτωση μη καταβολή των διοδίων θα πρέπει να είναι αναλογικά και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ε, και την ε, μη θελημένη παραβίαση της υποχρέωσης καταβολή των διοδίων σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει μια τέτοια περίπτωση να μπορεί κανείς να πληρώσει τα διόδια που του αναλογούν χωρίς επιβολή προστήμου και πιστεύω ότι η τεχνολογία προφανώς είναι το σημείο κλειδί για τα λειτουργικά συστήματα αλλά εκεί που δεν συμφωνώ είναι σε ό,τι αφορά την εισαγωγή της τεχνολογίας από το παράδειγμα 4 στο κείμενο της οδηγίας γιατί πιστεύω ότι οι σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας θα πρέπει να εκφράζονται το συντομότερο δυνατόν στην νομοθεσία. Άρα, σε αντίθεση με του προηγούμενου ομιλητέ, δεν πιστεύω ότι έχει νόημα να γίνει αυτό. Το θέμα της ευελιξία είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να έχουμε πράξεις κατά Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν νέε τεχνολογικές εξέλιξεις, να εκφράζονται πιο γρήγορα στο κείμενο χωρίς να χρησιμοποιούμε τη χρονοβόρα διαδικασία της συναπόφασης για να είμαστε λοιπόν πιο αποτελεσματικοί. Γιατί δεν πρόκειται αυτό να ωφελήσει αν καθυστερούμε τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την τροπολογία 3 και την τροπολογία 14. Δεν θα τι υποστηρίξω λοιπόν όσο έχουν στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και η πρόεδρο και ευχαριστούμε τον κύριο Φαμίλτερμπεργκ. Ο κύριο Νταλούντα. Σα ευχαριστώ πολύ χωρί μικρόφωνο. Ο κ. Δελούντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία αυτή. Και είμαι πεισμένο ότι η διαλειτουργικότητα θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο προκειμένου να επηρεαστεί και η κυκλοφορία και να χρησιμοποιούν να χρησιμοποιεί ο κόσμος άλλα μέσα μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να απλοποιηθεί η διαδικασία, να συμμετέχουν και πιο πολλά κράτη-μέλη και όχι μόνο τα κράτη-μέλη που έχουν διασυνοριακές περιοχές συνεργασίες όπως για παράδειγμα η Κοπεχάγη το Μάλμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει διαλειτουργικότητα με τέτοια συστήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλα συστήματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα και τη μεταφορά εμπορευμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Monsieur Madame Oui, euh, ε, δύο λεπτά. Στηρίζω πλήρως την πρόταση της Κομισιόν και του εισηγητή. ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της ε, διαλειτουργικότητας των, του εξοπλισμού διοδίων. Θυμάστε ότι όταν ε, μίλησα για τη δική μου έκθεση είχα πει ότι και η διαλειτουργικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δεν αρκούν τα λόγια, πρέπει να περνάμε και στις πράξεις, στα πρακτικά ζητήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτικής τιμολόγησης. Έχω κάποιες ερωτήσεις διευκρινιστικές να θέσω στον εισηγητή. Κύριε Σαλίνη, θα διευκρινίσετε την διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τηλεδιοδίων, ε, διευκρινίζοντας το ποιο ρόλο θα παίζει ο κάθε φορέας, ε, ο υπάροχη και οι διαχειριστές των συστημάτων. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογή δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και τα διόδια εντός πόλεων, τα αστικά διόδια. Ευχαριστώ. Κυρία Ντελμόντε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρότασή του. Νομίζω ότι η πρότασή του και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ενδιαφέρον ήγκη και πλέον η ώρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη διαλικουργικότητα των συστημάτων που θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τώρα, σχετικά με τις υπόλοιπες προτάσεις του εισηγητή, θα συμφωνήσω με αυτά που περιλαμβάνονται στην τροπολογία 1, για τους διαχειριστές των οδικών δικτύων έτσι ώστε να μην επιρρύπτονται υπερβολικά βάρη στους χρήστες. Και εγώ νομίζω ότι η τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει τον διάλογο ανάμεσα στα ευφυή e συστήματα οδήγησης και θα πρέπει μέσω της ψηφιοποίησης να διευκολύνουμε λύσεις οι οποίες να είναι ιδιαίτερως πρακτικές. Έτσι και αλλιώς οι προτάσεις μας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και εφικτές. Και τέλος, έχει σημασία να διευκολύνουμε την συζήτηση και την συμπερίληψη μάλλον των οδικών διοδίων στην ευρύτερη συζήτηση για τις μεταφορές στις διασυνοριακές περιοχές να μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές τα διόδια μπορεί να είναι ένα μέσο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε κάποιους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των συνεπειών αυτών, αποφεύγοντας τις τρευλώσεις της αγοράς. Ευχαριστώ κυρία Ντεμόντε για την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από τις συζητήσεις στην Επιτροπή μας υιοθετήσαμε και εμείς μια γνωμοδότηση για την διαλειτουργικότητα των τηλεοδιοδίων. Αντιλαμβάνομαι ότι το περιεχόμενο της είναι παρόμοιο με αυτό του κυρίου, της έκθεσης του κυρίου Σαλίνη. Να σας πω ποια είναι τα βασικά σημεία όμως της δικής μας έκθεσης και θα μιλήσω στη γλώσσα μου, στα λιθουανικά. Αυτή τη στιγμή πάνω από 20 κράτη-μέλη χρησιμοποιούν συστήματα τηλεοδιοδίων, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους όμως. Οπότε στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν να ενοποιηθούν, να εναρμονιστούν τα συστήματα τηλεδιοδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μειώσει ε, τις απώλειες εσόδων από μη πληρωμή διοδίων και επίσης θα αποφύγουμε και στρεβλώσεις ε, του ανταγωνισμού. Τα αυτοκίνητα θα έχουν συσκευές ε, εντός του ε, έχουν συσκευές εντός του οχήματος που πολύ συχνά είναι ακριβές θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τη χρήση άλλων συσκευών όπως ε, smartphones, ταμπλετών κλπ. Θα πρέπει όμως να επενδύσουμε σε λογισμικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες όλων των κρατών μελών. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε τις οργανωτικές πτυχές μας. Πρέπει να αποφύγουμε τα μονοπόλια, τη δημιουργία μονοπωλίων σε, σε αυτού του τον εξοπλισμό και θα πρέπει να συνδέσουμε τα συστήματά μας με το σύστημα UCARIS. Ε, οι επενδύσεις θα είναι μεγάλες. Και η Κομισιόν θα πρέπει να χρηματοδοτήσει ένα τμήμα, των, ε, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές μικρές εταιρείες και αυτοαπασχολούμενοι στον τομέα των μεταφορών Ενδεχομένω δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κόστο και υπάρχει λοιπόν και μια κοινωνική πτυχή. Θα πρέπει να εναρμονιστούν τα συστήματα ηλεκτρονικών διοδίων και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο. Θα πρέπει να επιτρέπει την χρήση υπάρχοντος εξοπλισμού, αλλά να είναι ανοιχτό και στην τεχνολογική καινοτομία. Τρίτον, θα πρέπει να δώσουμε βάρος στις κοινωνικές πτυχές. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur. Σας ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Τώρα να ακούσουμε τον εισηγητή. Μάλλον ευχαριστούμε τον εισηγητή από, το, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και να ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκθεση αυτή, τον κύριο Λουσβά. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατάρχά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Σαλήνη για το σχέδιο έκθεσης και για την γενικότερη υποστήριξη τη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς υποστηρίζεται το γενικότερο στόχο τη πρόταση της Επιτροπής, προώθηση της διαλειτουργικότητα των τηλεδιωτήων και επίσης υποστηρίζεται τη μεγάλη καινοτομία τη πρόταση, ένα νέο μηχανισμό ανταλλαγή πληροφοριών για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει καταβολή διωδίων από τους παραβάτες. Δεν θα αναφέρω τα θετικά, όπως και στις προηγούμενες εκθέσεις. Θα μιλήσω βέβαια για τις τροπολογίες που προβλέπουν ανταλλαγή πληροφοριών και χορήγηση πληροφοριών από τα εθνικά σημεία επαφής προς ε, τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι προωθεί την επιβολή του συστήματος. Σημειώνω ότι θέλετε να υπάρξει λίστα των τεχνολογιών και να συμπεριληφθεί στο διατακτικό της οδηγίας γιατί θεωρείται ότι είναι σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αλλάζει μόνο μέσω της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας Ακούσαμε ωστόσο διαφορετική άποψη του κυρίου Φαν Μίλτενμπρουχ και ακριβώς ο σκοπό της πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάζοντας σε παράρτημα τις τεχνολογίες αυτές είναι να γίνει πιο εύκολη και ευέλικτη και ταχεία η προσαρμογή και η ενημέρωση σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη σε ένα εύλογο χρονικό περιθώριο. Ε, Τίφεται λοιπόν θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα όπου η Επιτροπή διαφωνεί με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά την εξέρεξη των συστημάτων που χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ENPR, e αυτό με την αγνώριση της πινακίδας του οχήματος. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο εισηγητής προτείνεται προτείνει να διαγραφεί το σύστημα αυτό. Θεωρούμε ότι είναι σωστό για δύο λόγους. Καταρχάς, αν διαγραφεί το σύστημα αυτό, το σύστημα αυτό δεν θα ωφεληθεί από τη μεγάλη κοινοτομία της πρότασης που είναι η ανταλλαγή πληροφοριών για να εξασφαλίσουμε ότι οι χρήστες των υποδομών θα πληρώνουν τα αντίστοιχα διόδια. Και ξέρουμε ιδιαίτερως από τον διαχειριστή του συστήματος αυτού ότι υπάρχει ιδιαίτερα θέμα απάντηση ότι αφορά τη χρήση των συστημάτων. Χρήστες που δεν πληρώνουν δηλαδή. Και έτσι βλέπουμε όλα και πιο πολλά τέτοια συστήματα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία ένα τέτοιο σύστημα, θα δημιουργηθεί μια χώρα. Θα υπάρχει δυνατότητα ο κάθε πάροχο να παρέχει ευρωπαϊκέ λύσει για όλου του χρήστε είτε πρόκειται για εμπορικού χρήστε είτε για προσωπικού χρήστε. Εμεί θα θέλαμε λοιπόν να μπει στο πεδίο εφαρμογή ε, της ε, οδηγία του ENPR. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο το έθεσε ο κ. Σαλίνη. Το θέμα το θεσμικό, αν θέλετε, πέρα από την οδηγία. Διαπραγματευόμαστε με τα κρατημέλη την ε, την αναθεώρηση του συστήματος ETS, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόχων και των υπεύθυνων επιβολής ιδιωδίων και στις συζητήσεις μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και κυρίως με την νομική υπηρεσία προκύπτει ότι κάποιες διατάξεις της απόφασης της ETS ενδεχομένως να είναι στοιχεία αναπόσπαστα της ε, οδηγίας. Και στην περίπτωση αυτή δεν ε, μπορούν να εγκριθούν με πράξεις κατά εξουσιοδότηση και ενδεχομένως λοιπόν κάποια από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να μπουν στο διτακτικό της οδηγίας. Όπως είπε όμως και ο εισηγητής, είμαστε σε στενή επαφή και συζητάμε πισταμένως τα ζητήματα αυτά. Αυτά, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιζουά. Ο κύριος Σαλίνη έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους κοιόδης συγητές για τις παρατηρήσεις τις οποίες έκαναν. Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει η δυνατότητα να καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας γρήγορα. Τώρα για την κριτική που ασκήθηκε θα τα συζητήσουμε και θα τα δουλέψουμε περισσότερο. Ξεκινάω από την παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχικά εγώ είχα μια διαφορετική άποψη για τον ρόλο τον οποίο θα πρέπει να έχει το σύστημα ανάγνωσης ή ανείχνευσης των πινακίδων κυκλοφορίας. Στόχος, και το εξήγησα στους Κιώδης, δεν είναι να εξαιρέσουμε απόλυτα το βίντεο calling, αλλά να είναι ένα συνοδευτικό σύστημα ε, στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης είναι ένα μέσο το οποίο είναι σχετικά αξιόπιστο και σαν συνοδευτικό σύστημα είναι σαφές ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι τεχνικό εμάς το θέμα και θα το λύσουμε, δεν είναι πολιτικό θέμα. Έχουμε χώρο να δούμε τι θα κάνουμε σχετικά με τις υπόλοιπες παρατηρήσεις. Ε, πρέπει να βάλουμε τον κατάλογο των τεχνολογιών στο πλήρες σώμα της πρότασης και όχι σαν παράρτημα. Ε, νομίζω ότι η γνώμη μου είναι ότι μια τέτοια έκθεση είναι μια τεχνική οδογία και θα είναι σαν να βγάζουμε την κεντρική ουσία, αν θέλετε, αν βγάλουμε τον κατάλογο αυτό. Και αυτό θα μειώσει ακόμα και τη νομική ισχύ της πρότασης την οποία ετοιμάζουμε. Η απόφαση από τη φύση της είναι καλύτερα διαχρωμένη, αλλά δεν νομίζω ότι θα χάσουμε χρόνο σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να βιαστούμε. Έγινε επίσης αναφορά και στις αστικές μεταφορές. Εγώ στην παρούσα φάση έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε πλήρως τα θέματα ανάγνωσης και ανείχνευσης και τα ηλεκτρονικά διόδια. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να διακρίνουμε απόλυτα το, τα διόδια εκτός αστικών περιοχών και εντός των αστικών περιοχών. Ας ξεκινήσουμε με τα εκτός. Ε, υπάρχει τεράστιο κόστος λόγω ακριβώς της ε, έλλειψης ε, διάρθρωσης και διαλειτουργικότητας και αργότερα θα επανέλθουμε και στον αστικό χώρο. Σας ευχαριστώ κύριε Σαβίνη. Να θυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 20 Φεβρουαρίου, 12η μεσημβρινή. Θα συνεχίσουμε τώρα με τις δύο κατεξουσιοδότηση πράξεις για τα κοινά μέτρα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Θα ήθελα να ζητήσω την παρουσίαση λοιπόν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής της πρότασής της. Τέσσερα με πέντε λεπτά και μετά για να μας ενημερώσει για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις στον εισηγητή, τον υπεύθυνο με την βασική πράξη και θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι εφόσον το επιθυμούν. Αυτοί οι οποίοι αναχωρούν τις αιθούσεις παρακαλώ να το κάνουν σιωπηρά και να σεβαστούν τους συναδέλφους που παραμένουν. Λοιπόν, ε, όσοι θέλετε να πάρετε το λόγο, βγείτε από την αίθουσα. So, thank very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε να σας παρουσιάσω εν συντομία δύο κανονισμούς για την ε, κοινή διαχείριση της ασφάλειας στους αστροδρόμους. Ε, την πρώτη διαφάνεια, να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται, να σας πω ότι η ιδέα είναι να περιγράψουμε σε μια επίπεδο λεπτομέρειας ε, τι σιδηροδρομικές ασκήσεις και τι συνδρομικές δράσεις χρειάζονται για να υπάρχει ασφάλεια στους τεροδρόμους, Αλλά δεν ήθελα, δεν θέλαμε να μπούμε σε μεγάλο βαθμό λεπτομερίας και να γίνουν πολύ ε, συγκεκριμένες οι δράσεις αυτές. Και να είμαστε σαφείς, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο υπήρχε ήδη στο τέταρτο πακέτο για τους τεροδρόμους, αλλά φυσικά με τις αλλαγές στην νομοθετική διαδικασία ε, κατέστησαν σε κανονισμό Ρυθμίσει κατά εξουσιοδότηση λοιπόν. Η πρώτη που βλέπετε αφορά την διαχείριση των συστημάτων ασφαλείας τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τα συστήματα στρατομικών μεταφορών πρωτού πιστοποιηθούν. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε κάτι καινούριο εδώ. Μιλάμε για στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον τεχνικό πυλώνα του τέταρτου πακέτου για τους αεροδρόμους. Φυσικά η υπηρεσία στερεοδρόμων στη Βαλασιάν θα είναι η υπεύθυνη για τα πιστοποιητικά στερεοδρόμων σε τέτοιες ε, επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά λειτουργία διασυνοριακή. Και έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την αίρα ε, αντί για τις εθνικές ε, αρχές πιστοποίησης. Άρα θα πρέπει λοιπόν να αποτυπωθεί αυτός ο νέος ρόλος και αδράξαμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε το SCNSN e καθιστώντας σαφέστερες τις προδιαγραφές ασφαλείας για τις επιχειρήσεις. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση και σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, για παραδείγμα τη συμπεριφορά των υπαλλήλων. Σημαντική είναι η υπεύθυνη διαχείριση των συστημάτων ασφαλεία για την ασφάλεια των συνδρομικών μεταφορών. Και εδώ κοιτάμε ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με την ευθύνη των υπαλλήλων και των διαχειριστών ασφαλείας, πώς μπορούμε να μάθουμε από τα ατυχήματα που έχουν γίνει για να εξασφαλίζουμε ότι όχι μόνο θα ακολουθούνται οι κανόνες, αλλά έχουμε πραγματικά συστήματα τα οποία θα ενθαρρύνουν τον κόσμο να τρούν με υπεύθυνο τρόπο και πιο σημαντικό να μπορεί κανείς να μάθει και να ενταχθεί από περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η ασφάλεια που θέλαμε. Στο δεύτερο στοιχείο, εδώ αποτυπώνεται το ότι εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα των εθνικών κρατών, μελών και των εθνικών υπηρεσιών να εποπτεύουν την ασφάλεια. Είτε πρόκειται για πιστοποίηση εθνική, είτε πρόκειται για πιστοποίηση της ΕΡΑ. Προκειμένου λοιπόν να είναι η εποπτεία αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα εδώ και περνώντα στην επόμενη διαφάνεια τίφεται το θέμα το πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση που το πιστυπικό λειτουργίας έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και υπάρχει δεσνοριακή λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει λειτουργικότητα από όλες τις εθνικές υπηρεσίες για να υπάρχει κοινή εποπτεία. Αυτές είναι οι καινοτομίες, τα καινοτομικά στοιχεία, αν θέλετε, στο CSMR και πέραν αυτών. Βελτιώσαμε επευκαιρία και έκανα δύο ορισμούς. Και τέλος, τελική διαφάνεια για σήμερα, τελευταία διαφάνεια για σήμερα. Να σας πω πώς ε, πήγε η διαβούλευση. Να σας πω ότι καμία από τις CSMs αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα καινοτομικέ βασιζόμαστε σε συστάσεις ε, του περσινού Απριλίου από την υπηρεσία Δρόμων. Μετά από feedback πέρσι το καλοκαίρι έγιναν κάποια σχόλια. Δεν νομίζω σε κάθε περίπτωση ότι υπήρξε το οτιδήποτε ακαθόδες και διαφιλονικούμενο. Θα συγκεντρώσουμε λοιπόν όλα αυτά στις προτάσεις που έχετε μπροστά σας σήμερα. Αυτά και προφανώς αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση με χαρά να την απαντήσω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκινάμε την συζήτηση. Ο κ. Κράμερ ε, δεν είναι εδώ δυστυχώς. Ο κ. Μπάρ έχει το λόγο. Ε, να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση αυτό των πολυτεχνικών αυτών πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 για την κοινή μέθοδο ασφάλειας και κυρίως για το σημείο 2 για την εποπτεία. Να ρωτήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια πράγματα. Ποιο είναι ο συντονιστικός ρόλο της ΕΡΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει και αυτή ρόλο στο συντονισμό και ποια είναι η κοινή γλώσσα που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών. Σε δύο-τρία χρόνια θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε μία έκθεση για να αποφασίσουμε και να δούμε πώς έχει εξελιχθεί ο συντονισμός και να δούμε σε περίπτωση που κάποιος έχει αναλάβει την τον ηγετικό ρόλο ποιος ήταν αυτός. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αναφορές και τα σχόλια που πήρατε από τις εθνικές υπηρεσίες, τι έγινε σε ό,τι αφορά το ρόλο και την ενημέρωση και την ε, αλλαγή και προσαρμογή των εθνικών πιστοποιητικών. Και μία ερώτηση για τη διαδικασία. Ήσασταν ε, μαζί σε αυτές ε, τις ε, σύμφωτες διαδικασίας. Είχατε μήπως διαφορετική άποψη σε κάποιες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που α, υπάρξει ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα, ποιος ήταν ο ρόλος της ΕΡΑ, ποιος ήταν ο, λόγος, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις έρευνες, στις μετέπειτα. Η ΕΡΑ μπορεί να προβεί σε συστάσεις και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπάρ. Απάντηση Κομισιόν σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ο Βαντενκάπ, θέλατε το λόγο. Συζητώ συγγνώμη, δεν σας είδα. Σας ακούμε. Ε, Πρόεδρε, δεν με είδατε γιατί δεν είχα ζητήσει το λόγο. Αλλά μετά τη συζήτηση που άκουσα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του τεχνικών ερωτημάτων που έθεσε ο συνάδελφος ο κ. Μπαρ, θα ήθελα ως απλό κοινό νητό να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο να αυξήθηκε η ασφάλεια με τα μέτρα αυτά ή είναι πολύ νωρίς ακόμα. Καθότι θα πρέπει να φροντίσουμε και οι εκλογέ μας να παρακολουθούν λεπτό τι κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Άρα εγώ ρωτώ πολύ απλά, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα με την πρόταση αυτή. Merci pour cette grande... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βελτιώθηκαν τα πράγματα. Ε, παρακολουθούμε τις στατιστικές ασφάλειας ε, των κρατών μελών και το πανόραμα δεν είναι ίδιο σε όλες τις χώρες. Σε ορισμένες χώρες ε, τα πρώτα ποιότητα είναι, ε, ασφάλειας είναι πολύ ψηλά, ενώ σε άλλες ε, χώρες πιο χαμηλά, για λόγους ενδεχομένως συνολικού ύψους των επενδύσεων. Συνολικά βέβαια το συνδρομικό μας δίκτυο ε, είναι πιο ψηλό, ε, η ασφάλεια του είναι πιο ψηλή από τις οδικές μεταφορές ε, και γενικά είναι πολύ ασφαλές σύστημα. Η υπηρεσία ασφάλειας των σιδηροδρόμων παρακολουθεί, έχει ένα σύστημα παρακολούθησης των προβλημάτων που μπορεί να υποσκάψουν την ασφάλεια και προσπαθεί να βρει τρόπους να βελτιωθεί η ασφάλεια. Οι στατιστικές όμως δείχνουν ότι σε όλη την Ευρώπη συνολικά η ασφάλεια είναι σταθερή ή βελτιώνεται. Ιδιαίτερα ε, με περισσότερες επενδύσεις και πιο νέα τεχνολογία θα βρεθούμε σίγουρα σε πολύ καλή κατάσταση στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Θα ήθελα να χαιρετήσουμε την πρόοδο που έχει καταγραφεί στην έκθεση Κράμερ. Πρόκειται για θέματα πολύ σημαντικά για τις μεταφορές. Έχω και μία ερώτηση όμως. Πώς προετοιμάζονται τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή αυτών των καινούριων κανόνων. Πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, ε, έχοντας υπόψη τον ψηλό αριθμό ατυχημάτων που έχουν συμβεί για παράδειγμα στην Γαλλία με τρομακτικές καταστροφές ε, πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον τα προβλήματα αυτά πώς θα μειωθούν αυτά του, αυτού του τα ατυχήματα υψηλού προφίλ θα έλεγα σε ό,τι αφορά το τέταρτο συνδρομικό πακέτο τα οποία, το οποίο τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο ε, του επόμενου έτους να έχουν μεταγράψει στην Εθνική Νομοθεσία ε, μπορεί μάλιστα να φτάσει αυτή η προθεσμία μέχρι και τον Ιούνιο του 2020 αν τα κράτη, αν κάποιο κράτος μέλος το επιθυμεί, έχει αυτή τη δυνατότητα αρκεί να μας ειδοποιήσει μέχρι το τέλος του 2018. Είμαστε σε, σε στενές επαφές μέσω της Κανονιστικής Επιτροπής με όλα τα κράτη-μέλη και τους ε, ζητήσαμε ε, να έχουν ολοκληρώσει την μεταγραφή μέχρι τον Ιούνιο του 19. Δεν έχουμε ακόμα ε, νέα για το κατά πόσον έχουν προχωρήσει. Η υπηρεσία σιδηροδρόμων είναι σε επαφή με τις εθνικές αρχές έτσι ώστε να ερμηνευτεί με τον ίδιο τρόπο και να μεταγραφεί με τον ίδιο τρόπο αυτό το πακέτο. Ε, διοργανώσαμε πέρσι πολλές, πολλά συνέδρια και ημερίδες ε, σε διάφορα κράτη-μέλη και θα το κάνουμε και φέτος προκειμένου να δώσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα, να λύσουμε απορίες κλπ. Είναι λίγο νωρίς λοιπόν να γνωρίζουμε το κατά πόσον τα κράτη-μέλη έγκαιρα θα έχουν μεταγράψει το σύνολο αυτών των κανόνων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ατυχήματα. Πράγματι, πριν από τα Χριστούγεννα είχαμε ένα τραγικό ατύχημα στη Γαλλία. Κάθε ατύχημα είναι μια μεγάλη απώλεια. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ότι τέτοιου είδους ατυχήματα δεν σημαίνουν ότι πέφτει η ποιότητα της ασφάλειας. Το αντίθετο συμβαίνει. Βέβαια, είναι σαφές ότι με τις ισόπεδες διαβάσεις υπάρχει ένα ζήτημα Γίνονται πολλές επενδύσεις και πολλή δουλειά έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ισόπεδων διαβάσεων και περνώντας στα αυτόματα οχήματα, οχήματα χωρίς οδηγό κλπ. Ε, αναζητούμε καινούριους τρόπους για να αποφύγουμε ε, τέτοιου είδους ατυχήματα και αυτό θα το δούμε την επόμενη δεκαετία. Να απαντήσω και σε ερωτήσεις του κυρίου Μπάρ για τα ατυχήματα και το ρόλο της ε, υπηρεσία δρόμο και της Κομισιόν. Σύμφωνα με την οδηγία ασφάλειας, ο ρόλος ε, της διερεύνησης ατυχημάτων ε, είναι εθνικός, δηλαδή βαραίνει τα κράτη-μέλη. Αυτό γιατί το κείμενο είναι μια οδηγία. Η Εθνική Αρμόδια Αρχή Ασφάλειας ε, έχει λοιπόν την ευθύνη της διαρεύνησης τέτοιων ατυχημάτων και αναφέρει μετά στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδεοδρόμων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων δεν έχει ως καθήκον να κάνει συγκεκριμένες συστάσεις για συγκεκριμένα ατυχήματα. Τώρα, αν ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην αδειοδότηση, είτε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία είτε από Εθνική Υπηρεσία, τότε αυτό θα ήταν ένα σοβαρό ζήτημα και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά τα ίδια τα ατυχήματα και η διαρεύνησή του ε, είναι εθνική αρμοδιότητα. Merci σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις σας. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά τα τεχνικά, γιατί για μας έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το Κοινοβούλιο παρακολουθεί τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις με μεγάλο ενδιαφέρον και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο εξίσου με τους εμπειρογνώμονες των διαφόρων κρατών μελών. Θα πρέπει να έχουμε το ίδιο επίπεδο ενημέρωσης γιατί είμαστε συνομοθέτες. Σας ευχαριστώ και είστε καλοδεχούμενοι στην Επιτροπή μας. Συνάδελφοι, θα διακόψουμε τώρα. Θα βρεθούμε αύριο και θα ξεκινήσει η συνάντηση των συντονιστών στις 5.30.